Thank ψήφου λοιπόν ακολουθούν αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα αρχίσουμε με την έκθεση Lightfried σχετικά με μέτρα ασφαλείας για τις εναέριες μεταφορές. Η κυρία Οβίερ πρώτα, εάν είναι παρούσα. Έχετε το, το λόγο κυρία μου. Ε, δεν άκουσα το όνομά μου γιατί γίνεται πάρα πολύ θόρυβος μέσα στην αίθουσα του ημικυκλίου. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο έχει <clears throat> κατ' επανάληψη ζητήσει να ψηφιστεί σχετική νομοθεσία. Εγώ υποστήριξα την έγκριση του νομοθετήματος αφού είναι υπέρ όλων, της ασφάλειας όλων των επιβατών τα σχετικά τέλη να βασιστούν σε διαφανή κριτήρια. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ε, αποβούν εν τέλει υπέρ της ασφαλείας, δηλαδή να δαπανώνται για την ασφάλεια. Ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ, πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Όσοι εξημών επιθυμείτε να παραμείνετε, παρακαλώ να καθίσετε στα έδρανά σας. Και όσοι εξημών επιθυμείτε να ασχοληθείτε με άλλα, παρακαλώ εξέλθετε τις αιθούσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μέσα σε μια ήσυχη ατμόσφαιρα. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι σωστό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζουν το θέμα της διαφάνειας της χρηματοδότησης, της ασφάλειας των εναέριων μεταφορών. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ιδρύονται οργανισμοί για να ε, ασχοληθούν με το θέμα αυτό δεν είναι ο κατάλληλος. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από χρήματα για άλλα πράγματα, για να ενισχύσει την ελληνική οικονομία, για να αναπτύξει τη δική της η ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ η ίδρυση νέων εποπτικών οργανισμών στην ουσία σημαίνει κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων και δεν μπορεί να αποδώσει. Ο κύριος Λιμπεράτσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ε, μπόρεσα να υποστηρίξω, να ε, εγκρίνω με την ψήφο μου τον κανονισμό σχετικά με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και την πιστοποίηση αυτών εποφελία των χρηστών ε, αυτοκινήτων. Είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτύχουν δηλαδή καλύτερες τιμές. Άλλος κανείς, ρωτά ο πρόεδρος, θα ήθελε να εξηγήσει πώς ψήφισε για την έκθεση Lightfried. Αν όχι, μπορούμε να συνεχίσουμε με την έκθεση του κ. Σίμψον σχετικά με τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Ο κ. Κανσιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εχθές Καλώς πράξαμε που ολοκληρώσαμε την πρώτη ανάγνωση του ντοσιέ της ε, κωδικοποίησης. Ε, όμως υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που αφορά όλα τα δίκτυα νέου προγραμματισμού για την επόμενη δεκαετία. Αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν ορθολογικό τρόπο εντός της Ευρώπης, ώστε η διαλειτουργικότητα να είναι πραγματικά εφαρμόσιμη και εφαρμοστέα και στη διαδοχικά, επειδή έχουμε και την ε, αρνητική οικονομική κατάσταση, θα πρέπει να σκεφτούμε και την υλοποίηση αυτού του δικτύου ή τμήματος αυτού και όχι μόνο με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή αλλά να σκεφτούμε και μια διαφορετική διαδρομή, να μήπως μπορέσει η οικονομία να ανορθωθεί μέσω αυτού των δικτύων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πιο επίγον ακόμα να προσπαθήσουμε να δεσμευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς για την έκθεση Σίμψον. Όχι, σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την έκθεση Κυριλόφ. για τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής. Η κυρία Ομπύροβ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας υπέρ των τροπολογιών αυτής, ε, από αυτής εκθέσεως και αυτό διότι σέβομαι τους στόχους της δέσμης μέτρων οικονομικής ανάκαμψης που θα ενισχύσει τις επενδύσεις στις χώρες μέλη και στις περιφέρειες και θα έχει θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της οικονομίας και ιδίως όσον αφορά τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και τη δημιουργία απασχόλησης. Η απλοποίηση των κανόνων και διαδικασιών θα οδηγήσει στην επιτάχυνση της εφαρμογής και σε καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων. Ευχαριστώ, κυρία Μικουλενγκίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν υποστεί απώλειες τεράστιες κατά τη διάρκεια αυτής της οικονομικής κρίσης. Πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης είδαν ε, πτώση της οικονομίας τους μέχρι και 10%. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα, πρώην, τα παλιά και νέα κρατημέλη και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, ορθά τα διευθυντικά ταμεία που είναι ένα σημαντικό μέσο ε, που επιτρέπει να ξανασταθεί στα πόδια, τους η οικονομία των στα πόδια της οικονομία των κρατών μελών θα είναι πιο εύκολο για τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα αν χρησιμοποιηθούν σωστά τα διευθυντικά ταμεία. Ο, ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα μέσα για την ανάπτυξη των περιφερειών και για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που εδώ και ε, κάποιο χρόνο ε, ε, ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο τον κόσμο. Θα πρέπει να επιλοποιηθούν οι διαδικασίες ε, απελευθέρωσης των ε, κονδυλίων υπέρ των δικαιούχων των διαφόρων προγραμμάτων των λόγω ταμείων. Είμαστε υπέρ ενός επιπλέον ποσοστού προχρηματοδότησης για το 2010 για εκείνα τα κράτη-μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος για την έκθεση αυτή. Θα συνεχίσουμε με την έκθεση του κυρίου Σάιρ. Ο κύριος Αντωνιώτης έχει ζητήσει το λόγο για αυτή την έκθεση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξέφρασα την ψήφο μου υπέρ τη έκθεση του συναδέλφου Σάιερ, τον οποίο ήθελα να ευχαριστήσω για το εξαιρετικό αναλυτικό του έργο που έγινε με βάση τι ε, καινοτομίε τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και λόγω τη απλοποίηση τη νομοθετική διαδικασία ε, για τι ε, πράξει τι εξουσιοδοτημένε, νομίζω πω θα πρέπει αυτό να γίνεται με συγκεκριμένε και ξεκάθαρε Προποθέσει, ε, προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει ε, γνήσιος δημοκρατικός έλεγχος από πλευρά του Κοινοβούλιου. Θεωρώ πως θα, υπάρ... θα μπορέσει... Ε, μπορέσουν όλα αυτά να υλοποιηθούν στην πράξη για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα και ενδεχομένως να το διορθώσουμε αν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον που να θέλει να κάνει επεξήγηση ψήφου όσον αφορά την έκθεση ΣΑΙΡ. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα μας για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Η κυρία Θεοχάρους παρακαλώ. Που είναι και η μόνη εγγεγραμμένη. Η κυρία Θεοχάρους αν είναι εδώ. Κυρία Θεοχάρους παρακαλώ. Δεν είναι παρούσα η κυρία Θεοχάρους από ό,τι φαίνεται. Δεν βλέπω και κανέναν άλλο βουλευτή που να εκδηλώνει ενδιαφέρον να μιλήσει. Θα προχωρήσω στην έκθεση Βαντάλεν. Η κυρία Σαβισάρα. Η κυρία Σαβισάρ είναι απούσα από ό,τι φαίνεται. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην έκθεση Πάουλσεν. Πρώτος αγορητής που είχε ζητήσει το λόγο είναι ο κ. Καλινόφσκι. Κύριε Καλινόφσκι, παρακαλώ. Κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πιστεύω να μου δώσετε βέβαια δύο λεπτά μόνο και μόνο επειδή επιλύει ο προηγούμενο. Αλλά σε ένα λεπτό τέλο πάντων θα πω ότι υποστηρίζω την έκθεση που είναι σχετική με την προστασία και ευημερία των ζώων. Ωστόσο έχω ορισμένε επιφυλάξει σχετικά με το πώ νομοθετεί το Κοινοβούλιο και η Ένωση για το θέμα αυτό. Εγώ θα προτιμούσα μια επιστημονική θεμελίωση και λιγότερο συναισθηματική φόρτιση. Έχουμε νομοθεσία ήδη που σε πολλέ περιπτώσει δεν βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και οδηγεί έτσι τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε βαρύτατα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα. Είμαι πολύ δυσαρεστημένη για το γεγονός ότι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει συζητήσει αυτή την εβδομάδα με τις χώρες Μερκοσούρ, διακυβεύοντας έτσι το μέλλον των Ευρωπαίων παραγωγών και κυρίως σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέας και το ε, κρέας πουλερικών θα πρέπει να επιβληθούν οι ίδιες προδιαγραφές και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες όπως αυτές που επιβάλλονται στους εγχώριους παραγωγούς. Εάν δεν το κάνουμε αυτό πρόκειται πραγματικά για έσχος. Ευχαριστώ κύριε Μακίνες. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προστασία των ζώων είναι αδιαίρετη και πρέπει να ισχύει και παγκόσμια εναρμόνιση επομένω, Σε, ενώ, σε, ε, ε, ό,τι αφορά ναι, θέσπιση νέων προδιαγραφών α κάνουμε ένα διάλειμμα. Α φροντίσουμε πρώτα να υπάρξει μια ομοιόμορφη συμμόρφωση στους κανόνε αυτού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την παγκοσμιοποίηση. Α ενισχύσουμε τι προσπάθειέ μα, ούτω ώστε και οι εισαγωγέ από τρίτε χώρε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπακούν και να συμμορφώνονται στι ίδιε προδιαγραφέ όπω αυτέ που ισχύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, αυτό είναι δίκαιο του καταναλωτού να ε, ε, μπορεί να προμηθεύεται ασφαλή αλλά και ε, σωστά παρηγμένα προϊόντα. Άλλος κανείς για την, για την έκθεση αυτή. Κύριε Έκθεση του κύριου Λεφόλ. Η κυρία Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μην λησμονούμε ότι στα θεωρία βρίσκεται μια ομάδα επισκεπτών μου από την εκλογική μου περιφέρεια στην Ιρλανδία. Είναι σημαντικό οι πολίτες να ε, μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες του Κοινοβουλίου και βλέπετε ότι μας νεύουν φιλικά από τα θεωρία. Για την έκθεση αυτή είχαμε και έναν από τους Beatles εδώ που είπε ότι θα πρέπει να τρώμε λιγότερο κρέα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμω σε σχέση με τη γεωργία και την αλλαγή του κλίματο είναι να χρησιμοποιήσουμε την βέλτιστη τεχνολογία που διαθέτουμε για να μειώνουμε τι εκπομπέ που έρχονται από την αγροτική παραγωγή. Όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή ε, τροφίμων παγκοσμίω και θα το κάνουμε αυτό με λιγότερους πόρους, λιγότερο έδαφος, λιγότερο νερό και με την πίεση που ασκεί η κλιματική αλλαγή. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι η βέλτιστη δυνατή έρευνα που πρέπει να χρηματοδοτείται δημοσίως αλλά και με κοινοπραξίες του δυτικού και δημόσιου τομέα ώστε οι αγρότες να μπορούν να παράγουν τρόφιμα ασφαλή και με φιλικές προς το περιβάλλον ε, τεχνικές. Ευχαριστώ. Και χαιρετώ και εγώ την ομάδα επισκεπτών σας. Mm. Εσείς κύριε Γιάρα, τρία σύντομα σχόλια για την έκθεση αυτή. Πρώτα, η γεωργία δεν είναι το πρόβλημα, είναι περισσότερο η λύση του προβλήματος για την αλλαγή του κλίματος. Δεύτερο, έρευνα της αλλαγής του κλίματος. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, παρόλο που καμιά φορά τα μίδια λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. Για την έρευνα της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να δούμε και όλα τα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν από αυτήν, έστω και αν ορισμένα πηγαίνουν αντίθετα με αυτά που θεωρούμε ότι είναι σωστά. Να λαμβάνουμε λοιπόν μέτρα τα οποία να είναι επαρκή, κατάλληλα και επιστημονικά θεμελιωμένα και να ελέγχουμε και την αποτελεσματικότητά του στην οικονομία. Για παράδειγμα, για την οδηγία για προστασία του, έδαφου, του εδάφους που εν προκειμένου δεν, είναι, δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Άλλος κανείς για την έκθεση Λεφόλ. Όχι. Προχωρούμε. Στην ευεξήγηση ψήφου της έκθεσης Ντόρφμαν. Η κυρία Μαγκίνης και πάλι είναι γραμμένη. Ελπίζω να έχω εντυπωσιάσει όλους τους επισκέπτες μου δεν είναι συνθήσιμο να έχουμε τόσο πολύ χρόνο αγόρευση επεξηγήσει, αλλά επειδή με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα τη γεωργία. Περί τίνος πρόκειται εδώ, πώς θα καταφέρουμε να παραμείνουν οι αγρότες σε πολύ αντίξωες συνθήκες στην Ήπεθρο. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Γεωργοί είναι οι καλύτεροι διαχειριστές και του τοπίου και συντηρητές, αλλά χρειάζονται χρήματα για να επιβιώνουν στην Ήπεθρο τα οχτώ βιοφυσικά ε, κριτήρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω θα είναι υπερβολικά περιοριστικά όταν εγκριθούν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, τι διάφορε συνθήκε των εδαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ιρλανδία ανησυχούμε. Αν περάσουν αυτά τα κριτήρια και εφαρμοστούν στην περιοχή του Ατλαντικού, ε, θα υπάρχουν προβλήματα για τους αγρότες σε αυτές ακριβώς τις ακτές του Ατλαντικού. Παρακαλώ να το έχει υπόψη τη αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι είναι και η πιο φθηνή επιλογή που έχουμε και η καλύτερη να φροντίζουν οι αγρότες και τη γη και το τοπίο. Ας τους επιτρέψουμε να επιβιώνουν στις περιοχές τους λοιπόν. Ευχαριστώ. Χειροκροτούν οι επισκέπτες σας. Και τώρα πάμε στην έκθεση Ρέντερ Καστίγιο για τη νέα ψηφιακή ε, ατζέντα για την Ευρώπη. Η κυρία Αλφάνο είναι μοναδική ομιλήτρια. Ρέγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τη νέα ατζέντα της Ευρώπης για την ψηφιακή εποχή γιατί νομίζω ότι να εγγυωθούμε την προσιτή πρόσβαση στην ευρεία ζώνη για ολόκληρο τον πληθυσμό είναι στρατηγική προτεραιότητα για ολόκληρη την Ευρώπη. Διεύρυνση και της ελευθερίας έκφρασης των πολιτών σημαίνει αυτό με μεγαλύτερη δημοκρατικότητα και αυτό με οδηγεί στο να υπογραμμίσω πως η διάδοση του Εβραίου σφάσματος ολόκληρη την Ευρώπη έχει, είναι πολυδιάστατο θέμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Eurostat είπε ότι και όσον αφορά τη διάδοση του, του, του ίντερνετ υπάρχουν δύο διαφορετικές Ευρώπες. Η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και το Πορτογαλία αντιπροσωπεύουν τα κράτη που είναι λιγότερο ανεπτυγμένα ω ως προς το ίντερνετ. Ελευθερία τύπου ε, σε σχέση με το, για το 2009 η Ιταλία ε, αναφέρεται ως εμερικός ελεύθερη, τελευταία ευρωπαϊκή χώρα δίπλα με την Τουρκία. Η Ιταλική κυβέρνηση κατάφερε να απεμπλέξει τις επενδύσεις 800 εκατομμυρίων ευρώ που απευθύνονται για την ψηφιοποίηση της Ιταλίας και τελικά όντως ε, έχει καταστεί προτεραιότητα η ψηφιοποίηση της Ιταλίας. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτέ καταγγέλνουν πω το κόστο πρόσβαση είναι πολύ ψηλό στην Ιταλία, το ψηλότερο μάλιστα στην Ευρώπη. Κοιτάξτε να δείτε, την επόμενη φορά να ξέρετε, έχετε μόνο ένα λεπτό. Κανένα άλλο για την έκθεση αυτή, όχι. Έχουμε χρόνο να δώσουμε, να κάνουμε τις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση του Σάλα Σαλαφράγκα για τη Λατινική Αμερική. Ο κύριος Χίγκιν θέλει να πάρει το λόγο. Τουλάχιστον τον έχω στη λίστα μου εδώ. Όχι, δεν επιθυμεί. Οπότε δίνω το λόγο στον Καλύτερό μας ομιλητή σήμερα, την κυρία Μαγκίνε δηλαδή. Ευχαριστώ Πρόεδρε που με αναγνωρίζετε έτσι για να πω στους, ε, στους επισκέπτες μας ότι κανονικά ζητούμε να σιωπήσουν αλλά είμαστε πολύ επίκαιοι σήμερα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Το έχω ήδη αναφέρει αυτό και πιστεύω πως το Κοινοβούλιο δεν έχει ε, συνειδητοποιήσει στην έκθεση του Σαλαφράγκα τις επιπτώσεις της υποστήριξης αυτής της έκθεσης, πράγμα που δεν έπραξα εγώ. Πολύ με ανησυχεί η απόφαση να ξαναρχίσουν διμερείς ε, επαφές ε, με τις χώρες Μερκοσούρ. Καταρχήν, ε, ε, αυτά γίνονται γίνονται ενώ ταυτόχρονα γίνονται διαπραγματεύσει στον ΠΟΕ. Ε, γιατί πρέπει να κάνουμε διμερείς διαπραγματεύσεις. και επιπλέον, εάν ξεπουληθούμε όσον αφορά την γεωργία, και αυτά είναι οι δικές μου ανησυχίε. Ε, από ευρωπαϊκή ε, ε, άποψη θα είναι πολύ σημαντικέ οι επιπτώσει για την Ευρωπαϊκή Γεωργία αν φτάσουμε σε συμφωνίε σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Και πάλι ο ολόκληρο αγροτικό τομέα θα επηρεαστεί και κυρίω η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία. Γι' αυτό και καταψήφισα. Ευχαριστώ. Τελευταίο σημείο. Πριν να έρθει ο, πρόεδρο, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η ε, διάσκεψη κορυφής Ένωση Καναδάς. Ουγγίας είναι στον καταλογό μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το νερό είναι αγαθό για όλους. Δεν μπορεί να είναι μόνο για λίγους. Αυτό είναι μέσα στις αξίες της άλλης, σε σχέση με την τροπολογία 10 που ήταν αντίθετη, αντίθετη με οποιαδήποτε απόπειρα ιδιωτικοποίησης των εταιριών διανομής του νερού που αποτελεί τμήμα της συνολικής οικονομικής ε, συμφωνίας και είμαστε δεσμευμένοι μαζί με τους Καναδούς για να, να εμποδίσουμε την ιδιωτικοποίηση του νερού. Εμείς ε, θελήσαμε να επιψηφίσουμε το κείμενο γιατί αντιπροσωπεύει τις αξίες μας, αυτές μας οδηγούν στο να επιβεβαιώσουμε την ε, ε, φύση του του κοινού αγαθού για το νερό. Έχουμε συγκεντρώσει και υπογραφές με ένα δημόσιο δημοψήφισμα κατά το ιδιωτικοποίηση του νερού της διανομής του νερού και συγκεντρώνουμε ακόμα τέτοιες υπογραφές σε μεγάλο αριθμό. Συνάδελφοι, μόλις έλαβα την πληροφορία πως θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση όσον αφορά τον αντιπρόεδρο, την άφηξη του